Μαλεσίας. Η κυρία Βάιλερ για 1,5 λεπτό πρώτη για να παρουσιάσει το ψήφισμα. Εφαρμογή ποινών ξυλοδαρμού. Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι. Είναι εντυπωσιακή χώρα η Μολεσία, μια χώρα με παλιές παραδόσεις, με πολιτιστικό πλούτο ως, μέλος της, ε, ως μέλη της Επιτροπής ΑΖΕΑΝ είχαμε την ευκαιρία πολλές φορές να παρακολουθήσουμε τις ταχείες και εντυπωσιακές εξελίξεις στο κράτος αυτό. Και η οικονομική ρόμη της Μαλαισίας που ε, αυξάνεται διαρκώς δείχνει την ε, ταχύτατη πορεία της Μαλαισίας με μια οικονομική ανάπτυξη η οποία την εντάσσει στις πρώτες δέκα σε ανάπτυξη χώρες στον κόσμο. Θα ήθελα λοιπόν γι' αυτό να σημειώσω και ευχαριστώ επί τη ευκαιρία όσους συνυπέγραψαν μαζί μου και το ψήφισμα πώς είναι δυνατόν στη σύγχρονη εποχή το σύγχρονο αυτοκράτος η Μαλαισία να εφαρμόζει ακόμη μία ε, απαρχαιωμένη μορφή ε, κολασμού, μια μορφή που ανήκει για τη Μαλαισία στην απεικιοκρατική εποχή, ενώ για μας ακόμη σηματοδοτεί τον Μεσαίωνα. Πιστεύουμε ότι θα πρέπει πολύ γρήγορα να αλλάξει αυτή η κατάσταση. Με πολύ μεγάλη χαρά βλέπουμε ότι εκδόθηκε ο χάρτης, ε, η χάρτα των κρατών ΑΣΕΑΝ, που με απερίφραστα λόγια και παραθέτω στα αγγλικά, αναφέρεται ότι στόχος ουσιώδης των ε, χωρών ΑΣΕΑΝ είναι η προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας. Στα κράτη αυτά βέβαια έχει ενταχθεί και η Μαλαισία, άρα είναι στρατευμένη και δεσμευμένη να υιοθετήσει και τις δημοκρατικές αρχές, αλλά αυτό σημαίνει και κράτος δικαίου με οικουμενικέ αρχές. Άρα οποτεδήποτε επισκεφτόμαστε τη Μαλαισία και τα άλλα κράτη του ΑΣΕΑΝ και πιστεύω θα μπορέσει να το ενισχύσει αυτό και το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πρέπει να υπογραμμίζουμε αυτή τη διάσταση. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Σάκε, για ένα μισή λεπτό. Πρόεδρε, κυρίε και κύριοι, η μορφή αυτή του ξυλοδαρμού με με κάλαμο, ε, του ραφτισμού δηλαδή, είναι ένα μέσον το οποίο γνωρίζει ακόμα δυστυχώς η Μαλαισία. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο ενισχύεται, εφαρμόζεται πολύ συχνά εις βάρος μεταναστών και αποτελεί παραβίαση της, ε, των οικουμενικών δικαιωμάτων και των σχετικών διακηρύξεων ε, που καταδικάζουν κάθε μορφή σωματικού κολασμού δεν υπάρχει δυνατότητα ε, για τα θύματα των σχετικών καταδικών ούτε για ε, αντίδραση με ένδικα μέσα στις σχετικές αποφάσεις ούτε καν της υποστήριξη από δικηγόρο. Γι' αυτό απευθύνουμε έκκληση να σταματήσει αυτή η υπόθεση, αυτό το σύστημα ε, σωματικού κολασμού και ταυτόχρονα να στηρίζουμε τους δικηγόρους και τις οργανώσεις των θυμάτων που αγωνίζονται για την κατάργηση αυτού του μέσου. Θα πρέπει η κατάργηση της ε, σχετικής νομοθεσίας να προχωρήσει το χέτερο δυνατό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Σάκε. Η κυρία λοχμπιλα Πρόεδρε, ευχαριστώ. Με το ψήφισμα αυτό καταδικάζουμε τις, ε, τις ποινές ξυλοδαρμού, ραβδισμού, αντίστοιχων σωματικών κυρώσεων και κολασμού στις, ε, στη Μαλαισία που αποτελούν τα ταπεινωτικές ε, ποινές, όπως τις εννοεί και η Σύμβαση κατά των βασανιστήριων για την ε, θέτει τέρμα στα βασανιστήρια. Η πρακτική λοιπόν εφαρμογή αυτών των ε, βασανιστήριων και των ποινών, των βάναυσων στη Μαλαισία συνεχίζεται δυστυχώς και εξομοιώνεται με βασανιστήρια. Για 66 τουλάχιστον αδικήματα προβλέπει η Μαλαισιανή νομοθεσία αυτή τη βάναυση μεταχείριση και ιδιαιτέρως ε, από πέρυσι έχει ε, εισαχθεί ως μέτρο εις βάρος λαθρομεταναστών που παράνομα δηλαδή έχουν μπει στο κράτος ή εις βάρος εξαρτημένων από ναρκωτικές ουσίες, ναρκωμανών. Είναι πολύ μεγάλος αριθμός δηλαδή των ανθρώπων που πλήττονται, από αυτή, που κινδυνεύουν από αυτή την ε, βάναυση ταπεινωτική προσβλητική της αξιοπρέπειας του ανθρώπου πίνει και καλούμε την Μαλαισιανή κυβέρνηση να την αποσύρει από το νομοθετικό του σώμα. Είναι μέλο του Συμβουλίου για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα η Μαλαισία τη ΑΣΤΑΝ και όπω είπε και η συνάδελφο νωρίτερα, απαγορεύονται οι, ε, οι, σωματικοί, οι κολλασμοί, ε, ο ξυλοδαρμό και αντίστοιχα μέσα ω είδη βασανιστήριων από τη σχετική σύμβαση, την οποία καλούμε τη Μαλαισία να εφαρμόσει το δυνατό. Ευχαριστώ πολύ κυρία Λόχμπιλ. Ο συνάδελφος Τάνοκ, πρόεδρε, ε, η Μαλαισία φαίνεται ότι στρέφεται προς μια Ισλαμική μορφή διακυβέρνησης. Είναι κρίμα αυτό και ανησυχητικό γιατί θα μπορούσε να ήταν σύμμαχος και τέρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης η Μαλαισία. Κάποιες ε, έννοιες του δυτικού πολιτισμού φαίνεται ότι χάνονται από τη Μαλαισία. Ε, στον πληθυσμό ο, η πλειοψηφία είναι μουσουλμάνοι και τέτοιου είδους τιμωρίες είναι ε, συνήθις στο Ισλάμ και στις χώρες που εφαρμόζεται ο νόμος της Σαρία και μάλιστα είναι και ελαφριά ποινή τελικά διότι στη Σιγκαπούρη λόγου χάριν ε, ε, Υπάρχει και εκεί, ε, υπάρχει και η ποινή του ξυλοδαρμού και σε άλλες γειτονικέ χώρες γίνεται το ίδιο. Βεβαίως οι σωματικές ποινές στη Δύση απαγορεύονται αλλά τελικά δεν ξέρω αν υπό το διεθνές δίκαιο είναι παράνομη, απαγορεύεται η ποινή του ξυλοδαρμού όπως λέγεται στο ψήφισμα. Ο κύριος Πόσελτ, πρόεδρε, άμα αγαπάει κάποιος κάποιον τότε έχει και συγκεκριμένες απαιτήσεις. Ε, όταν πρόκειται λοιπόν για χώρες με τις οποίες είμαστε στενά συνδεδεμένοι τότε έχουμε διαφορετική στάση από ότι σε σχέση με άλλες δικτατορίες σε άλλα μέρη του κόσμου η Μαλαισία είναι φίλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης βεβαίως έχει ένα σύνταγμα το οποίο μπορεί να επιτρέπει ορισμένα πράγματα που δεν μας αρέσουν εμάς. Ο ξυλοδαρμός αγαπητέ συνάδελφε Τάνοκ στην Μαλαισία δεν εισήχθη από τον νόμο της Σαρία αλλά από τους Βρετανούς απεικιοκράτες από εκεί και πέρα κάποιες μεταρρυθμίσεις και αλλαγές θα έπρεπε να γίνουν και σίγουρα θα πρέπει να ζητήσουμε να γίνουν και αλλαγέ για τέτοιου είδους ποινές οι οποίες είναι ενάντια στο διεθνές δίκαιο. Η Μαλαισία όμως πρέπει να παραμείνει όπως ήταν και παλιά στενός εταίρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να τους βοηθήσουμε να ξεπεράσουν αυτή τη βαρβαρική ποινή ευχαριστώ πολύ ο κύριος Τάνο ξαναζητά το λόγο να ρωτήσω κάτι τον κύριο Πόσελτ. Τον σέβομαι απόλυτα και βεβαίω εγώ δεν γνωρίζω το διεθνές δίκαιο αλλά δεν νομίζω ότι υπάρχει απόδειξη ή κανένα αποδεικτικό στοιχείο που να λέει ότι ο ξυλοδαρμό αυτού του είδους με βέργα ή το μαστίγο ο ραβδισμός αυτός απαγορεύεται από το διεθνές δίκαιο. Και μάλιστα στη Μαλαισία λένε ήδη ότι θα μπορούσε αυτός ο ραβδισμός να θεωρηθεί βασανιστήριο αλλά που δεν είναι λόγο μπορώ να θεωρήσω ότι ο ραβδισμός είναι βασανιστήριο. Ο κύριος Πόσελτ ε, ναι ναι Θεωρώ ότι ήταν ερώτηση αυτή και θα ήθελα να απαντήσω ότι βεβαίως είναι βασανιστήριο η τιμωρία αυτή και βεβαίως είναι ενάντια στα ανθρώπινα δικαιώματα και στο διεθνές δίκαιο. Βεβαίως. Ευχαριστώ κύριε Πόσελτ. Ωραία λοιπόν. Η κυρία Μπερζιά, μισή λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η Μαλαισία είναι μία από τις χώρες με τις οποίες ε, η πρόσφατη συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση φαίνεται ως κάτι θετικό. Υπάρχει και οικονομική πτυχή αλλά και η κοινωνική πτυχή αυτής της βοήθειας σε θέματα εκπαιδευτικά ε, γυναικών ή στήριξη των πιο ευάλωτων πληθυσμών. Δυστυχώ, ε, σε θέματα δημοκρατία και ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η κατάσταση δεν είναι καθόλου ειδηλιακή. Ε, τα μηνύματα που λαμβάνουμε από τη Μαλαισία είναι ανησυχητικά και ιδού η απόδειξη. Παρόλο που η Μαλαισία έχει προσυπογράψει πολλές διεθνείς συμβάσεις όπως την Οικουμενική ε, Συνθήκη Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, δυστυχώς δεν θέλει να υπογράψει την Διεθνή συνθήκη κατά των βασανισμών. Είναι από τις χώρες που εφαρμόζεται θανατική ποινή η Μαλαισία και μάλιστα η θανατική ποινή είναι υποχρεωτική σε περίπτωση λαθρεμπορίων ναρκωτικών. Πολύ συχνά εφαρμόζονται σωματικές τιμωρίες και προς όλες τις κατευθύνσεις ε, έναντι πάντων ε, κατά ανδρών, γυναικών, ακόμη και παιδιών και γυναικών που έχουν ε, κατηγορηθεί για εξωσυζυγικές σχέσεις ή κατά μαθητών που είναι απίθαρτη στα μαθήματα. Μερικές φορές μάλιστα αυτές οι ποινές εφαρμόζονται με τη συνενοχή των γιατρών που καταπατούν το διοντολογικό τους κώδικα και που συνεφέρουν τους τιμωρημένους μόλις λιποθυμήσουν. Δυστυχώς ε, ε, είναι πολλές αυτές οι παραβιάσεις. Πάνω από 60 είχαμε τέτοιες περιπτώσεις και από το 2002 όταν δημιουργήθηκε αυτή, όταν δημιουργήθηκε αυτό το, αυτό το έγκλημα, χιλιάδες άνθρωποι υπέστησαν λόγω λάθρα μετανάστευσης παράνομη εισόδου στη χώρα τον ξυλοδαρμό. Θα πρέπει λοιπόν να δρέψουμε τους καρπούς αυτής της συνεργασίας με τη Μαλαισία χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε μέσα έχουμε στη διάθεσή μας και αντιπιθώ πάνω απ' όλα για να βοηθήσουμε τη Μαλαισία να προχωρήσει προς το τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Συνάδελφε Βερζιά για θα ήθελα να πω ότι δεν ε, θα ήθελα οι ομιλητές να ξεπεράσουν, ξεπερνούν το χρόνο ομιλίας τους κατά παραπάνω από ένα τρίτο ε, παρόλο που διαπνέουμε από ένα χριστουγεννιάτικο πνεύμα παρόλα αυτά έτσι πρέπει να προχωρήσουμε διότι διαφορετικά δεν θα τελειώσουμε ποτέ ο κύριος Πρέντα Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα καταρχήν να σας μεταφέρω κάποια στοιχεία από μια πρόσφατη μελέτη του τελευταίου μήνα από τη Διεθνή Αμνηστία. Τουλάχιστον 10.000 άνθρωποι και 6.000 πρόσφυγες υφίστανται την ποινή του ραβδισμού κάθε χρόνο. Και τέτοιοι ραβδισμοί λαμβάνουν χώρα στη φυλακή. Και δυστυχώς, όπως είπε ο κύριος Τάνοκ, η Μαλαισία δεν είναι η μοναδική χώρα που εφαρμόζει αυτή την αναχρονιστική σωματική τιμωρία. Μιλούμε εδώ και για τη Σιγκαπούρη, αλλά αυτό που με ανησυχεί κυρίως για τη Μαλαισία είναι ότι εκεί έχουμε πολύ μεγαλύτερο αριθμό εγκλημάτων που τιμωρούνται με ραβδισμό. 66 αδικήματα στη Μαλαισία τιμωρούνται με ραβδισμό ενώ είναι 30 μόνο τα σχετικά εγκλήματα στην Σιγκαπούρη. Δεν μιλούμε μόνο για σεξουαλικά εγκλήματα αλλά και για ε, χρήση ναρκωτικών ή παραβίαση της νομοθεσίας περί μετανάστευσης που επισύρουν τέτοια ποινή. Θα πρέπει να παροτρύνουμε την Μαλαισία να προσυπογράψει τις διεθνείς συμβάσεις για την απαγόρευση του βασανισμού. Ο κύριος δεν μπόρεσε να έρθει. Έχει τη συγγνώμη η κυρία Γιατενακή. Για ένα μισή λεπτό. Πρόεδρε, είναι πολύ σημαντικό το ψήφισμα αυτό του Κοινοβουλίου. Έρχεται την κατάλληλη στιγμή. Έχουμε χιλιάδε ανθρώπων που πέφτουν θύματα του ραβδισμού στη Μαλαισία κάθε χρόνο. Πρόκειται για μια απάνθρωπη μορφή, μια βάνευση μορφή τιμωρία που θα πρέπει να καταργηθεί σε ολόκληρο τον κόσμο. Είναι μια μορφή βασανιστηρίου. Μία μουσουλμάνα γυναίκα ε, ε, ραβδίστηκε πέρυσι στην Μαλαισία όπου εφαρμόζεται ο κανόνας της ε, Σαρία και με βάση τις, με τα στοιχεία της Amnesty International και ο λόγος για τον οποίο υπέστη το ραβδισμό αυτό ήταν ότι την έπιασε να πίνει μπύρα. Κυρίες και κύριοι, είναι μια μορφή απάνθρωπης τιμωρίας ο ραβδισμός. Την καλούμε λοιπόν να την καταργήσει και ταυτόχρονα την καλούμε να ακυρώσει το πρωτόκολλο των ΗΠΑ για, την, ε, για τα βασανιστήρια, την απαγόρευση των βασανιστήριων, καθώς και το αντίστοιχο πρωτόκολλο για τα ανθρώπινα και πολιτικά δικαιώματα. Ευχαριστώ πολύ την κυρία Γιατεράκη. Και τώρα ο κύριος Σούμπρο, παρακαλώ, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ με ιδιαίτερη ικανοποίηση. Διαπιστώνουμε ότι τα τελευταία χρόνια η Μαλαισία αναπτύσσεται οικονομικά με ραγδαίου ρυθμούς. Δυστυχώ όμω πρέπει να λάβουμε υπόψη και τη μελέτη τη Διεθνούς Αμνηστία που μιλά για την εφαρμογή τη ποινή ραβδισμού στη Μαλαισία. Φυσικά είναι πολύ σοβαρή αυτή η ποινή και πολλέ φορέ επιβάλλεται για πολύ μικρά δικήματα έως και παραπτώματα. Και ιδιαίτερα εφαρμόζεται έναντι λαθρομεταναστών που μπαίνουν στο έδαφος της Μαλαισίας χωρίς ταξιδιωτικά έγγραφα χωρίς διαβατήριο και εφαρμόζεται αυτή η αυστηρή πίνη. Μερικές φορές βέβαια ε, είναι και παραδοσιακός ο λόγος, πολιτιστικός για, την, για τον οποίο επιβάλλεται ο ραβδισμός και είναι συνήθως ε, η εφαρμογή του Ισλαμικού νόμου, της Σαρία, που οδηγεί στην ε, πίνη του ραβδισμού. Μάλιστα είχαμε την περίπτωση της ε, μουσουλμάνας γυναίκας το 2009 που υπέστη την ποινή του ραβδισμού μόνο και μόνο επειδή βρέθηκε να καταναλώνει μπύρα. Είναι απαράδεκτο αυτό. Το λόγο έχει ο κύριος Πάσκα για 1,5 λεπτό. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ο Ισλαμικός ε, Εθνικός Νόμος, η Σαρία, που εφαρμόζεται σε πολλές μουσουλμανικές χώρες προβλέπει σωματικές ποινές για την διάπραξη αδικημάτων. Είχαμε την περίπτωση της γυναίκας, της γυναίκας που υπέστηθε την ποινή μόνο και μόνο επειδή ε, κατανάλωσε μπύρα. Και είχαμε και την περίπτωση ενός διατάγματος ε, που επέβαλε την ποινή ε, μαστίγωσης, ε, ραβδισμού έναντι μιας γυναίκας μητέρας τριών παιδιών και μάλιστα τελικά έγινε μετατροπή της ποινής σε τρεις μήνες καταναγκαστικά έργα. Είχαμε πολλές περιπτώσεις Ε, τέτοιων ποινών και μάλιστα είναι άδικη η επιβολή αυτής, αυτής της ποινής και διαφορετικά επιδικάζεται εις βάρος ε, γυναικών και εις βάρος ανδρών. Για, την ίδια, για το ίδιο αδίκημα, για παράδειγμα, σε έναν άνδρα επιβλήθηκε μόνο ε, έξι χτυπήματα. Ο Υφυπουργό Παιδεία δικαιολόγησε την ποινή του ραβδισμού έναντι παιδιών στα σχολεία με το επιχείρημα ότι είναι ποινή που βελτιώνει την κατάσταση στα σχολεία θα πρέπει να ενημερώνει το επιθεωρητή του σχολείου και, τα παιδιά, ε, και οι γονείς των παιδιών απλώς. Θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε λοιπόν κάθε διπλωματική με διαβλό προκειμένου να βοηθήσουμε αυτές τις χώρες να καταργήσουν αυτές τις αμεσαιωνικές και αναχρονιστικές ποινές. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα το λόγο έχει ο κύριος Σόνι. Φυσικά καταδικάζουμε τη χρήση ποινή ε, ραβδισμού ή οποιασδήποτε σωματική ποινή και απάνθρωπη ε, μεταχείριση. Δεν μπορεί να εφαρμόζει εθνικό δίκαιο που προβλέπει ποινή ραβδισμού για 66 αδικήματα και μάλιστα άσχετα μεταξύ τους. Ο ραβδισμός με βάση διεθνείς συνθήκες χαρακτηρίζεται ως ε, σωματικός βασανισμός. Μάλιστα η Διεθνής Αμνηστία ε, λέει ότι η ποινή αυτή εφαρμόζεται κυρίως εις βάρος λαθρομεταναστών. Θα πρέπει ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση να χρησιμοποιήσει πολύ πιο αποτελεσματικά μέσα για να υπερασπίσει τα ανθρώπινα δικαιώματα και να λάβει περισσότερες πρωτοβουλίες για να καταπολεμηθεί η χρήση τέτοιων ποινών στον κόσμο. Τα θεμελιώδη δικαιώματα και η προστασία τους ε, είναι σημαντικός όρος που θα πρέπει να απαιτεί την τηρήση του Ευρωπαϊκή Ένωση για περαιτέρω αναπτυξιακή και οικονομική συνεργασία με χώρες όπως η Μαλαισία. Σας ευχαριστώ για ένα λεπτό. Το λόγο έχει ο κύριος Τσαρνέτσκι. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, η Μαλαισία είναι οικονομικός τίγρης, είναι πολύ ανεπτυγμένη οικονομικά χώρα, που μάλιστα αποτελεί υπόδειγμα για την ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ασίας. Αυτός ο τίγρης όμως έχει ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Και το πρόβλημα του τίγρη είναι ακριβώς αυτή η ποινή του ραβδισμού. Θα μπορούσαμε να πούμε για την ε, τήρηση και το σεβασμό κάποιων ε, πολιτιστικών ιδιαιτεροτήτων. Εμείς οι Ευρωπαίοι είμαστε πολύ ευαίσθητοι σε ό,τι αφορά αυτή, αυτό το σεβασμό των πολιτιστικών ιδιαιτεροτήτων και θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί όταν επιβάλλουμε τα δικά μας μοντέλα στον κόσμο. Αλλά στην περίπτωση αυτή μιλούμε για θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα. Αυτά τα θεμελιώδη δικαιώματα δεν γνωρίζουν σύνορα, δεν γνωρίζουν θρησκείες ούτε εθνότητες. Θα πρέπει λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση πολύ πιο στεναρά να ταχθεί υπέρ τη προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τη ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Γιατί πραγματικά η εφαρμογή τη ποινή του ραβδισμού παραβιάζει αυτή την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Σα ευχαριστώ. Η κυρία Μακοβέη, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η χρήση σωματική ε, τιμωρία ε, αποτελεί παραβίαση ανθρωπίνη αξιοπρέπεια. Είναι είναι παραβίαση της απαγόρευσης των βασανιστήριων αλλά και της απαγόρευσης μειωτικής ή απαξιωτικής μεταχείρισης ή συμπεριφοράς ο ραβδισμός. Και όμως είναι χιλιάδες οι άνθρωποι που υποφέρουν από αυτή την απαξιωτική συμπεριφορά και την τιμωρία η ε, στη Μαλαισία. Οι εκθέσεις δεν αναφέρουν ότι μερικές φορές φτάνουν μέχρι λιποθυμίας οι ραβδισμοί αυτοί. Οι δε αξιωματικοί οι οποίοι τις επιβάλλουν δέχονται και δωροδοκία ακόμη προκειμένου να την ε, μειώσουν, να μειώσουν την έντασή της. Απαιτείνω λοιπόν έκκληση προς την Επιτροπή και το Συμβούλιο αλλά και προς την κυβέρνηση της Μαλαισίας να επιβάλλει αμέσως μορατόριο στην ποινή του ραβδισμού και να προχωρήσει στην κατάργηση της σχετικής νομοθεσίας. Πρέπει να σταματήσει ο ξυλοδερμός, η, άσκηση σωματικής βίας, ο ραβδισμός και κάθε μορφή βασανιστήριων. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Είναι λυπηρό το ότι στη Μαλαισία ο ραβδισμός έχει φτάσει σε τέτοιες ακρότητες. Οι αρχές της Μαλαισίας χρησιμοποιούν ένα ανυπόστατο επιχείρημα, ένα βάσιμο επιχείρημα, ότι, είναι, ότι δεν είναι παράνομος ο ραπτισμός και ότι έχει στόχο τον παραδειγματισμό. Φαίνεται βέβαια από τις ε, εκθέσεις ότι πέφτουν θύματα κάθε χρόνο αυτού του φαινομένου, αυτής της ε, πάθρωπης μεταχείρισης, ε, τουλάχιστον 10.000 κρατούμενοι στις φυλακές και 6.000 λαθρομετανάστες. Είναι αδύνατον ε, στην ε, Μαλαισία να περιμένει κανείς ότι θα έχει μία δίκη με ισότιμες συνθήκες, μία μερόλεπτη δίκη, ούτε καν δικαίωμα στη διερμηνία δεν έχουν. Ευχαριστώ πολύ λέει ο Πρόεδρος και τώρα περνάμε στη δικασία του Καρστιάε με τον κύριο Ρέιπορτ πρώτα. Ε, Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Η ποινή του ραβδισμού και μάλιστα όταν ο κατηγορούμενος είναι δεμένος σε ένα στήλο και έχει έκθετη την πλάτη του που τη χτυπούν με ένα ραβδί με μια βέργα, είναι πραγματικά μια εξευθυλιστική σωματική ποινή και μάλιστα στη Μαλαισία έχει φτάσει τις διαστάσεις ε, επιδημίας. Ε, οι μαλαισιακές αρχές θεωρούν ότι οι σωματικές ε, ποινές, οι σωματικές τιμωρίες είναι ένας ε, αποτελεσματικός τρόπος για τον παραδειγματισμό των εγκληματιών και τον περιορισμό της εγκληματικότητας. Δεν θα πρέπει όμω να συνεχίσουμε την αναπτυξιακή βοήθεια και την οικονομική βοήθεια σε μια χώρα που εφαρμόζει τέτοιε ποινέ. Θα πρέπει να σταματήσει επιτέλου η χώρα αυτή να τι επιβάλλει. Μπορούμε λοιπόν να ζητήσουμε, να απαιτήσουμε από τι αρχέ τη Μαλαισία να σταματήσουν αμέσως την ε, επιδίκαση και την εφαρμογή τέτοιων ποινών και ε, νόμο και στην πράξη. ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η μαστίγωση εφαρμόζεται στη Μαλαισία από το 19ο αιώνα όταν η Μεγάλη Βρετανία επίκησε τα εδάφια εκείνα. Το τελευταίο καιρό μάλιστα η Μαλαισία έχει διευρύνει το κατάλογο αδικημάτων που επισύρουν την ποινή της μαστίγωσης και τα εγκλήματα αυτά έχουν φτάσει στα 66 τώρα. Και μάλιστα οι άνθρωποι που τιμωρούνται με, τις, με την ποινή του ραδισμού κρατούνται σε φυλακές χωρίς καμία ενημέρωση για το χρόνο επιβολής. Ε, η Διεθνή Αμνηστία μας ενημερώνει ότι 10.000 ε, τέτοιες αποφάσεις έχουν εκδοθεί και μάλιστα το 60% επιβάλλονται σε λαθρομετανάστες που εξαιτία άγνοιας γλώσσας δεν γνωρίζουν ε, καν το περιεχόμενο της απόφασης. Θα πρέπει λοιπόν να, να στην στενή μας συνεργασία με την Μαλαισία εδώ τα τελευταία 8 χρόνια να το θίξουμε αυτό. Από στις δημοσιονομικές προοπτικές 2007-2013 έχουν προβλεφθεί 17 εκατομμύρια ευρώ για την βοήθεια προς τη Μαλαισία. Είναι σημαντική πρόκληση να ζητήσουμε από τον εταίρο μας να κυρώσει την σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για την κατάργηση των βασανιστήριων και θα πρέπει επίσης να υποδηλώσουμε στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ αυτή την κατάρτιση πρακτική της Μαλαισίας. Η κυρία Κρέτσου, για ένα λεπτό. Κυρία. Πρόεδρε, πάνω από 10.000 πολίτες ε, υφίσταται την τιμωρία αυτή στην Μαλαισία του χρόνου ε, με, ε, γιατί στην ποινή αυτή υπόκειται τουλάχιστον 66 αδικήματα. Επεκτάθηκε η, η γκάμα τα τελευταία χρόνια. Επιπλέον οι κρατούμενοι οι οποίοι υπόκεινται στην τιμωρία αυτή δεν ενημερώνονται, δεν έχουν σωστή διερμηνία κτλ. Θα ήθελα λοιπόν να καλέσω όλους να, να συνεχίσουν την πίεση για να καταργηθεί η πίνη αυτή. Ε, θέλουμε ε, δίκαιες δίκαιες στη Μαλαισία και σωστή μεταχείριση των κρατουμένων ή των λαθρομεταναστών. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Ο Επίτροπος Πίμπαλξ έχει το λόγο. Πρόεδρε, αξιότιμοι ευρωβουλευτές, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καταδικάζει την χρήση την ύπαρξη σωματικών ποινών. Είναι αντίθετο με τα, αντίθετη μια τέτοια τιμωρία με τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν ανταποκρίνεται στις αρχές μας η, πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τρίτες χώρες δεν μπορεί να η, μην διαπιστώσει μέσα στα πλαίσια αυτών πολιτικών δεν μπορούμε να διαπιστώσουμε κάποια τέτοια πράγματα που συμβαίνουν σε τρίτες χώρες. Εμείς θα θέλαμε, συμφωνούμε με το ψήφισμα αυτό, αλλά θα θέλαμε να διευρυνθεί το ψήφισμα αυτό σε όλες τις χώρες όπου υφίσταται ακόμη η ποινή αυτή. Και βεβαίω πολύ σωστά κάνατε και ε, αναβασχοληθήκατε με το θέμα αυτό και πολύ αναφέρθηκαν βεβαίως στην ε, συνθήκη των Ηνωμένων Εθνών για τα βασανιστήρια. Θυμηθείτε και τις συζητήσεις που έγιναν το Φεβρουάριο του 2009. Την περασμένη εβδομάδα σε ένα σεμινάριο των Ηνωμένων Εθνών με βάση την ημέρα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ε, η Μαλαισία ε, εκλήθη να προσπογράψει τη Σύμβαση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και ιδιαίτερα την ε, ε, Σύμβαση κατά των βασανιστήριων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση στη Μαλαισία θα αρχίσει διαπραγματεύσεις για μια συμφωνία εταιρική σχέσης η οποία θα περιλαμβάνει και διατάξεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Όταν τεθούν σε συμφωνία λοιπόν αυτές οι συμφωνίες θα αποτελούν μια στέρεα και τυποποιημένη βάση για διάλογο και νομικό διάλογο ακόμη με τη Μαλαισία για τα ανθρώπινα δικαιώματα και ταυτόχρονα θα αρχίσουμε να εγείρουμε το ζήτημα αυτό με τις αρχές της Μαλαισίας. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε, κύριε Πίβαλ. Έξι προτάσεις ψηφισμάτων έχουν 7 Β7-0709-2010 των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών.